Καλημέρα σε όλες και όλους. Morning Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό περιλαμβάνει και εσάς κύριε Βαντεργάμπ. So, be... Αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήλθατε. Έχουμε πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε. Δύο ημέρες συνεδρίασης της Επιτροπής μας που είναι υπερφορτωμένες σε επίπεδο ημερήσιας διάταξης. Έχουμε πλήρη λοιπόν ατζέντα. Πρωί, απόγευμα, πρωί, απόγευμα. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν το ταχύτερο δυνατό. Στι 11 και 10 θα γίνει ψηφοφορία. Θα γίνουν οι ψηφοφορίε, τέσσερι ψηφοφορίες. Και θα έχουμε τότε μεγαλύτερη προσέλευση συναδέλφων που είναι πρόθυμοι <clears throat> να περάσουν στην ψηφοφορία για τα σημεία αυτά. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τη χρήση του χρόνου. Ξεκινάμε λοιπόν με τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Καταρχήν έχουμε την έγκριση των πρακτικών. <clears throat> Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης, 9 Φεβρουαρίου, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα αν δεν υπάρχει αντίρρηση μέχρι το τέλος της αυριανής ημέρας. Και πάμε κατευθείαν στο σημείο 4. Έχουμε την κοινή συνάντηση, συνεδρίαση με την Νομική Επιτροπή για το πρόγραμμα εργασίας 2014-2020, κοινή συνεδρίαση όπως είπα μεταξύ Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Ευχαριστούμε την κυρία Εύελιν Βέγνερ που είναι παρούσα. Εκπροσωπούσα την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Έχουμε τον κύριο Κλέης από τη δική μας Επιτροπή και τον κύριο Μπερλιγκουέρ από την Νομική Επιτροπή και θα ακούσουμε τις απόψεις τους για τις τροπολογίες σε σχέση με ένα κανονισμό ο οποίος θεσπίζει το πρόγραμμα δικαιοσύνης για το 2014-2020. Έχουμε λοιπόν <clears throat> την εφαρμογή του άρθρου 51 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ επιτροπών. Έχουν κατατεθεί 79 τροπολογίες και προβλέπεται να ψηφιστούν στις 27 Νοεμβρίου. Θέλω λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Ρέγνερ που είναι αντιπρόεδρος της Νομικής Επιτροπής και μετά <clears throat> θα δώσω το λόγο στους ε, συνεισηγητές, τον κύριο Κλέης και στον κύριο Μπέρλιγκουερ. Κυρία Ρέγνερ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Λόμπε Αγγιλάρ. Εξ ονόματος της Νομικής Επιτροπής θέλω να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με την έκθεση αυτή. Καταρχήν, υπάρχει μια μακρά παράδοση σε σχέση με τη θαυμάσια συνεργασία μεταξύ της ε, Νομικής Επιτροπής και επί της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών για τα θέματα αυτά. Ανατρέχοντας το παρελθόν στην έναρξη αυτής της νομοθετικής περίοδου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για τη συνεργασία μας για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και άλλες εκθέσεις, οι οποίες εκπονήθηκαν στα πλαίσια μιας θαυμάσιας συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη επίσης για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης που να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία αναγνώριση. Η έκθεση λοιπόν αυτή για το πρόγραμμα δικαιοσύνης 2014-2020 είναι ο διάδοχος του προγράμματος που υπάρχει ήδη για την δικαιοσύνη και την πρόληψη της εγκληματικότητας και είναι μια ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Θα ήθελα να αναφέρω μόνο το θέμα της χρηματοδότησης, γιατί είναι ένα από τα κέρια θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η Κομισιόν προτείνει 472 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση, αλλά ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι ο τελικός. Δεν, είτε, δεν έχει πει κανείς τον τελικό λόγο, διότι όλα αυτά εξαρτώνται από τις διαπραγματεύσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα σε σχέση με, τον πολυ, με τις πολυετείς δημοσιονομικές προοπτικές. Κατά τα άλλα μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε και αποτελεσματική νομοθεσία, αλλά χρειαζόμαστε και τους απαραίτητους δημοσιονομικούς πόρους για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Και όπως είπε και ο πρόεδρος Λόπες Αγγιλάρ, έχουμε 79 τροπολογίες. των εισηγητών που έχουν εκπονηθεί μεταξύ του κύριου Κλέης και του κύριου Μπέλιγκερ. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι η τελική ψηφοφορία θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου και πάλι σε μια κοινή συνεδρίαση της Νομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών και ελπίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει θα είναι επικοδομητικό στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τους δύο εισηγητές. Θα ξεκινήσουμε με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, τον κύριο Μπέρλιγκουερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προετοιμασία της έκθεσης στο συγκεκριμένο θέμα έγινε τους τελευταίους μήνες. Είχα στενή συνεργασία με τον κύριο Κράιες και νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα συγκλίνον αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα υπόδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στην Επιτροπή Γιούρη και ανάμεσα στα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, κάτι το οποίο μας βοήθησε πολύ να προχωρήσουμε. Ακούσαμε αρκετές προτάσεις από πλευράς των ενδιαφερομένων. Είχαμε συνεχή επαφή, διαρκή επαφή και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι καταφέραμε χτες να καταλήξουμε. Θα σταθώ σε πέντε σημεία σύντομα. Το πρώτο αφορά την παρουσία των ναρκωτικών σε αυτό το πρόγραμμα. Όχι στο συνολικότερο πρόγραμμα της Ένωσης, αλλά στο συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα για την δικαιοσύνη. Έχουν κατατεθεί τροπολογίες 43, 51, 52 μέχρι 68 έγινε συζήτηση αν πράγματι το θέμα των ναρκωτικών θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ως έχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, για την δικαιοσύνη. Όχι τόσο τα θέματα της πρόληψης, όχι τόσο τα θέματα της υγείας που δεν αφορούν τις δύο αυτές επιτροπές. Κατατέθηκαν λοιπόν αρκετές τροπολογίες Επί τη βάση αυτών των τροπολογιών προσπαθήσαμε να επεξεργαστούμε το κείμενο για να τις λάβουμε υπόψη. Είχαμε, θα έλεγα, απορρίψει την άποψη του Συμβουλίου, το οποίο έλεγε ότι δεν πρέπει τα ναρκωτικά να συμπεριληφθούν. Αυτό είχε ζητήσει το Συμβούλιο, να φύγει το θέμα των ναρκωτικών, λέγοντας ότι θα έπρεπε να συζητηθεί σε διαφορετικά πεδία συζήτησης. Εν πάση περιπτώσει θα υπάρξουν συγκεκριμένα προγράμματα για την υγεία και για την πρόληψη και εμείς ε, ε, θα αφήσουμε ανοιχτή τη συζήτηση και στη συνέχεια θα επανέλθουμε. Σαν κοινοβούλιο εμείς θα πρέπει νομίζω να μείνουμε ανοιχτοί. Σχετικά τώρα με τους δείκτες, οι τροπολογίες 87, 92 και 19 έχουν σαν στόχο να εντάξουν τους δείκτες τους οποίους είχαμε ήδη εμείς προτείνει στην αρχική μας πρόταση. Είχαμε προτείνει επίσης σαν τρίτο θέμα μία τροπολογία, την 33, σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, είδαμε ότι η πρόθεσή τους είναι να μην υπάρχουν κατεξουσιοδότης πράξεις εδώ, αλλά εκτελεστικές πράξεις με διαβουλευτική διαδικασία, με διαβούλευση. Εμείς νομίζω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε το θέμα αυτό ανοιχτό σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Σχετικά τώρα με αυτούς οι οποίοι θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα, το θέμα είναι ευαίσθητο θα έλεγα. Ήρθαμε σε επαφή στενή με τους ενδιαφερομένους. Είχαμε και τις παρεμβάσεις των Προέδρων Λένε και Λόπες, ο συνάδελφος Κλέης και εγώ όπως και όλοι οι σκιώδεις εισηγητές, ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας, ζήτησαν να ακολουθηθεί η αρχική λύση. Η καταγραφή αυτών οι οποίοι ωφελούνται θα είναι πιο χρήσιμη και στην προκαταπτική αναφορά στο πρόγραμμα και όχι τόσο στο τελικό κείμενο του προγράμματος. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο παραδείγματος επιλέξαμε τρία θεσμικά όργανα, αλλά η διατύπωση είναι τέτοια που επιτρέπει φυσικά και ε, σε άλλα όργανα να τύχουν των συγκεκριμένων οικονομικών προβλέψεων. Λοιπόν, εμείς καταφέραμε να ξεπεράσουμε τελικά λοιπόν τις πιθανές διαφορές το θέμα δεν είναι αν θα υπάρξει ένας κατάλογος των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το θέμα είναι αν θα περιλαμβάνεται ο κατάλογος αυτός η καταγραφή των οργάνων που θα τύχουν οικονομική στήριξη στην αιτιολογική σκέψη ή στο ε, ε, επίσημο κείμενο. Λοιπόν, είναι θέμα πρακτικό και όχι τόσο θα έλεγα λειτουργικό και ουσιαστικό. Με τον συνάδελφο Κλάι συζητήσαμε και την τροπολογία για τα δικαιώματα των παιδιών, των ανηλίκων. Υπήρξαν αρκετά θέματα προς συζήτηση. Υπάρχει ο κίνδυνος εμείς να καταλήξουμε σε ένα κείμενο στο πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη, το οποίο να είναι εξαντλητικά αναλυτικό. Πάντως η πρότασή συγκεκριμένη είναι αποδεκτή και θα καταλήξουμε σε μια λύση πιο συγκεκριμένη και πιο περιληπτική των προτάσεων που έχουν γίνει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κλάης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βεβαίω υπάρχει κίνδυνο να επαναληφθώ, αλλά και εγώ θα ήθελα ε, να αναφερθώ στην ε, καλή συνεργασία που είχαμε και με όλου του συναδέλφου και στην έκθεση, αλλά και με του κοιόδη συζητητέ. Όταν ε, για πρώτη φορά συζητήσαμε σε αυτή την επιτροπή το κείμενο αυτής της έκθεσης, όταν ετέθη στη διάθεσή μας, είχαμε ήδη καταλήξει σε μια συνένεση, έτσι νόμιζα, ακούσαμε και τις διάφορες πολιτικές ομάδες και τώρα εκπλήσωμε από τον αριθμό των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Έχουμε περίπου 80 τροπολογίες. Όπως και να έχει, νομίζω ότι μπορούμε να τις ομοδοποιήσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Υπάρχει μεγάλος αριθμός τροπολογιών για τα ναρκωτικά, άλλες ε, τροπολογίες ε, για την, ε, για όχι μόνο κατασταλτική δράση ε, και προσέγγιση, τις οποίες θεωρώ αρκετά αξιόλογε, και μετά άλλες τροπολογίες που ε, συμπεριλαμβάνουν κάποια στοιχεία πρόληψης και όχι μόνο καταστολής. Και αυτά τα στηρίζουμε. Υπάρχουν όμως και άλλες τροπολογίες που προσπαθούν να μας βάλουν σε μια διαφορετική συζήτηση. Γιατί τίθεται και θέμα ορολογίας που θέλουμε να εισαγάγουμε ε, και για το αν θα κάνω μια διάκριση μεταξύ μαλακών και σκληρών ναρκωτικών. Ε, και εγώ ειλικρινά, βεβαίω είμαι πάντα διαδεθειμένο να κάνω τέτοια συζήτηση. Φοβάμαι όμω ότι ε, αυτή η συζήτηση βρίσκεται εκτό του πλαισίου αυτή τη έκθεση. Ανοίγεται μια συζήτηση που δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ και δεν πρέπει να κάνουμε εδώ όταν συζητάμε το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη 2014-2020. Υπάρχουν ε, για κάποιε τροπολογίε, όπω ανέφερε ο συνάδελφο, ε, που αναφέρονται στην προστασία των ε, δικαιωμάτων των παιδιών και εκεί μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό, πιστεύω. Άλλες τροπολογίες επί του κειμένου, επί της διατύπωσης, δεν είναι απαραίτητες για μένα, ε, για ζητήματα που καθορίζονται και στις συνθήκες ή για την διασυνορία και συνεργασία, ε, όπου θέλει κάποιος να προσθέσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Βεβαίως μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοιες προτάσεις και εμείς αναγνωρίζουμε προβλήματα που υπάρχουν με τα δικαιώματα των παιδιών. Ε, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, της εμπορίας ανθρώπων, ε, ιδίως ό,τι αφορά τους ανηλίκους, αλλά κατά βάση ένα τέτοιο κείμενο πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση της ε, ως το μεγαλύτερης ευκρίνειας και εφαρμοστικότητας και μετά τέτοιε παρατηρήσεις μπορούμε να τις βάλουμε στις αιτιολογικές σκέψεις αντί για το ίδιο διατακτικό. Όπως είπα και προηγουμένως, ο κ. Μπελιγκουάρη και εγώ συμφωνούμε με αυτούς τους δείκτε ε, για την μέτρηση των αποτελεσμάτων για να καταστεί το έργο μας ε, πιο ε, σαφές. Λάβαμε και τροπολογίε από αυτού από τις ε, πολιτικές ομάδες. και προτείνω αυτό αυτέ τι προτάσεις να τι περιλάβουμε στι συμβαστικές μας προτάσεις. Όπως είπε και ο Μπερλιγκουέρ, για τι καταξιδιώτε πράξει ε, έναντι τη ε, έναντι της δυνατότητας ε, ύπαρξης εκτελεστικών πράξεων. νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε ως το μεγαλύτερο αντίκτυπο κατά την την επιλογή του νομοθετικού πλαίσιου. Ας ακούσουμε τώρα τις αντιδράσεις των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Okay, we thank you for your... Εντάξει, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας <clears throat> και για την παρουσίαση μια σύνοψη των τροπολογιών. Η Προεδρία τώρα αν ήθελε να λάβει το λόγο σε αυτή τη φάση. Πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη. Βλέπω να ζητάτε το λόγο. Εάν όμως <clears throat> η Προεδρία του Συμβουλίου θέλει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις, θα ήθελα να τους ζητήσω να το κάνουν εν συντομία. Παρακαλώ. <clears throat> Στο 8 Ιουνίου το Συμβούλιο κατέληξε σε μια γενική μερική προσέγγιση. Αυτή η γενική αλλά και μερική προσέγγιση δεν συμπεριλαμβάνει τα αριθμητικά ποσά όπως ε, συζητούνται στην ε, ομάδα για τις δημοσιονομικές προοπτικές από την ομάδα των φίλων της Προεδρίας και δεν έχουμε λοιπόν περιλάβει όλα αυτά τα στοιχεία σε αυτή την προσέγγιση. Κάποια κράτη-μέλη μέσα στο Συμβούλιο πρότειναν να υπάρξει κάποια διαίρεση μεταξύ του προγράμματος για την υγεία <clears throat> και του προγράμματος για την αστυνομία και τα υπόλοιπα να πάνε στο πρόγραμμα των ε, νομικών θεμάτων. Η νομική βάση της, ε, του κανονισμού θα παραμείνει όπως έχει και οι δράσεις οι οποίες θα καλυφθούν από αυτόν τον κανονισμό θα παρουσιαστούν από την ε, Προεδρία επισήμως και σε ό,τι αφορά τη γενική αυτού του του θέματος. Αυτό καλύπτεται από την οριζόντια ομάδα εργασίας DRAX, η οποία θα καλύψει τα κενά στις δράσεις οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί ακόμα και θα εξασφαλίσει την ε, αποφυγή ενδεχομένων επικαλύψεων. Επί της ουσίας τώρα του κανονισμού σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, η γενική μερική προσέγγιση συμπεριλαμβάνει στους στόχους της την υποστήριξη στην εκπαίδευση των δικαστικών και στους ειδικού στόχους συμπεριλαμβάνει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, των δικαστικών συστημάτων και τη συνεργασία της με, με τη χρήση ε, τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και σε διαμεθοριακό επίπεδο διαλειτουργικότητος και την πρόσβαση στο πρόγραμμα αυτό βάσει της γενικής μερικής προσέγγισης του Συμβουλίου θα προσανατολίστε και σε σώματα και φορείς που είναι κερδοσκοπικούς χαρακτήρας αλλά μόνο για δραστηριότητες που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, η Κομισιόν μπορεί να συνεργαστεί με διεθνείς φορείς επί τη βάση των ε, προδιαγραφών που θεσπίζονται στα ετήσια προγράμματα και η πρόσβαση στα προγράμματα αυτή, αυτά είναι ανοιχτή και για διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του προγράμματος επί τη βάση του δημοσιονομικού κανονισμού. Σε σχέση με τους ενδείκτες, το Συμβούλιο έχει καθορίσει τα συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων και η Προεδρία του Συμβουλίου σε αυτή τη φάση θέλει να συνεχίσει τις τεχνικές συναντήσεις επεξεργασίας με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να υπάρξει εναρμόνιση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στη γενική μερική προσέγγιση του Συμβουλίου. Η κυρία Μισού για την Κομισιόν θέλει να κάνει κάποιες παρατήρησεις, εν συντομία. Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ. Καλημέρα. Ακούσαμε τις ε, εξηγήσει ό,τι αφορά τα κύρια ζητήματα των τροπολογιών. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό. Απλώς, στο τέλος των συζητήσεων πρέπει να έχουμε προτάσεις και προγράμματα που θα είναι πολύ ξεκάθαρα, πολύ πρακτικά στην υλοποίησή τους, να να προσθέτουν κάτι στην πολιτική και να βοηθούν και τους δικαιούχους. Ε, για όλα αυτά πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη ισορροπία. Στις τροπολογίες που εξέτασα υπάρχουν βέβαια όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε μετά από συζητήσεις. Όμως πρέπει να δούμε σφαιρικά για όλα τα προγράμματα της Επιτροπής, ε, αν δηλαδή αυτά τα προγράμματα ή άλλα προγράμματα που έχουν εξεταστεί, ε, μπορούν να συμπληρώσουν το ένα το άλλο. Τελικά λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε αρκετά ζητήματα που είναι οριζόντια. Ε, κάποια από αυτά, όπως είπατε, είναι η καταξιδότηση πράξης, τα ναρκωτικά, αλλά ε, τελικά θα πρέπει να έχουμε ένα πραξης τα ναρκωτικα αλλα τελικα θα πρεπει να εχουμε ενα απλο στην εφαρμογή του πρόγραμμα. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Ας δώσουμε το λόγο στα μέλη τώρα. Τα μέλη που θέλουν να παρέμβουν. Ας ξεκινήσουμε από την Αντιπρόεδρο, κυρία Γκόγκς. Thank you very much. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Υπάρχουν ε, πολλές ε, παρόμοιες ε, τροπολογίες μεταξύ της Γιούρη και της Λίμπε που θα μας δώσουν ένα ισχυρό υλικό στο τέλος. Κάποια καλά στοιχεία. Η προληπτική δικαιοσύνη. Αυτή η έννοια έχει εισαχθεί και στις δύο επιτροπές. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να διατηρηθεί ως ιδέα. Μετά, η στήριξη της συγκριτικής ανάλυσης ενωσιακού και διεθνούς δικαίου είναι σημαντικό θέμα γιατί έχουμε περιορισμένες γνώσεις ε, σε ό,τι αφορά το, το δίκαιο του άλλου και έτσι πρέπει να υπάρχει ένας ε, βαθμός εμπιστοσύνης γιατί υπάρχει το θέμα του διοικητικού άχθους ε, που επανέρχεται σε όλες τις προτάσεις. Κάτι που έχει αναφερθεί πολλές φορές είναι τα δικαιώματα των παιδιών. Πρέπει να διατηρηθεί εδώ μια ισορροπία και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση των διακρίσεων. <coughs> Πρέπει να δούμε πώς θα το καλύψουμε αυτό το θέμα εδώ ή σε άλλα προγράμματα δικαιωμάτων και ηθαγένειας. Και και η ηλεκτρονική μάθηση βεβαίω είναι πολύ σημαντικό θέμα. Εμείς ε, παλεύουμε για ένα ανεξάρτητο ε, σύστημα δικαιοσύνης που καταπολεμά ε, τις πρακτικές διακρίσεων και παρέχει και διασφαλίζει ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Επικεντρωνόμαστε και στην πρόσβαση στα δικαιώματα, δηλαδή πρόσβαση σε δικηγόρο και το καθεξής. Ε, και να εξετάσουμε και τι συμβαίνει με αυτά τα, τα θρηστικά δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν. Ε, εμείς εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ε, λόγο ετησίως ό,τι συμβαίνει με τα προγράμματα, σε ό,τι αφορά την απλούστευση των διαδικασιών, γεωγραφική ισορροπία, συνδρομή προς τα κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν ακόμα. Κάποιες πιο προβληματικές τροπολογίες αφορούν συγκεκριμένε οργανώσει που είναι δύσκολο και επικίνδυνο μάλλον το να αναφέρουμε συγκεκριμένου οργανισμού εδώ. Ε, γιατί είναι και το θέμα των λόμπι. Επομένω, καλό θα ήταν να αποφύγουμε να κατανομάσουμε οργανισμού. Απλώ να περιγράφουμε τι είδου οργανισμών ε, πρέπει να είναι δικαιούχοι. Αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο. και υπήρχαν κάποιε τροπολογίε ότι πρέπει να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση για του δικαιούχου με το να περιορίσουμε το μερίδιο ε, τη χρηματοδότησή του σε σχέση με τον ετήσιο προπολογισμό. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο συγκεκριμένοι, αλλά θα υπάρξουν και επόμενε συζητήσει ε, με του εκπροσώπου τη Επιτροπή και του Συμβουλίου και σίγουρα ε, θα καταλήξουμε σε μια δυνατή πρόταση. Ο κύριος Βαντερκάμπ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές ε, για τις σκληρές προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι τώρα. Έχω την εντύπωση, Πρόεδρε, ότι η σημασία του προγράμματος δικαιοσύνης 2014-2020 ε, παραγνωρίζεται λίγο σε αυτό το κοινοβούλιο. Ε, τα μεγάλα παιδιά της ε, ε, των περιφερειών και της γεωργίας καθορίζουν μάλλον τη συζήτηση ότι φορά το πολιτισμό νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα και προς εσάς και προς τη συνάδελφο Ρέχνερ. Αν το ύψος, αν προσέχετε τι συμβαίνει με το ύψος του προπολογισμού σε αυτές τις διαπραγματεύσεις γιατί συμβαίνουν, λαμβάνουν χώρα διάφορες ε, μυστικές και λιγότερο μυστικές ε, συζητήσει, αλλά πρέπει ε, και εμείς να είμαστε θεματοφύλακε του προπολογισμού. Και θέλω να με ρημνήσετε ούτως ώστε ο προπολογισμό μας θα διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα και ή δυνατόν θα αυξηθεί κιόλας. Αυτό σας το έχω ήδη πει. Ναι, και εγώ αυτό προσπαθώ, κύριε Βαντερκάμπ. Ωραία ε, και θα σας ε, στηρίξω και θα σας ε, επικρίνω αν αυτό είναι δυνατόν βεβαίως. Ε, και για τον κύριο Κλάς θα πρέπει να, τον ξυπνήσω λίγο γιατί ο αριθμός των τροπολογιών είναι πολύ καλός. Στην Επιτροπή Ρέτζη υπήρχαν 220 τροπολογίες. Ας μην παραπονιέται ο κύριος Κλάς λοιπόν για τον αριθμό των τροπολογιών. Μια χαρά θα τα βρούμε. Βεβαίω το θέμα είναι πότε μπορούμε να περιμένουμε τι ε, συμβιβαστικέ τροπολογίε, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ε, για κάποια κείμενα βεβαίω δεν υπάρχει πρόβλημα, ιδίω για τα παιδιά, ας για τα δικαιώματα των, παιδιών. Μπορούμε να περιορίσουμε τον ε, αριθμό των τροπολογιών με την εξέβρεση συμβιβαστικών τροπολογιών. Ε, κύριε Πρόεδρε, το ΕΛΚ είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με τις τροπολογίες της κυρίας Βρίσπεκ ε, της Άλντε έχει υποβάλει τροπολογίες που απλοποιούν τα πράγματα και είμαστε θετικά διακείμενοι. Πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί με τέτοιου είδους προγράμματα για να μην αυξάνεται το διοικητικό άχθος και η γραφειοκρατία και ε, για τις τροπολογίες κυρίας Γκρίσβεκ θα ήθελα και τις ε, αντιδράσεις των ε, εισηγητών, αν δηλαδή μπορούν να τι αποδεχθούν. Τώρα, για το ζήτημα της κατάρτισης των δικαστών, έχω δύο ερωτήματα εδώ. Αφενός, έχουν υποβληθεί τροπολογίες ε, για την διεύρυνση της έννοιας των δικαστών και για, που να περιλαμβάνει πλέον και άλλο δικαστικό προσωπικό. Εμείς συμφωνούμε με αυτό. Ε, η γνώση σε αυτό το τομέα στην Ολλανδία είναι πολύ περιορισμένη, γι' αυτό θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας ε, σε αυτό και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα με την κυρία Γκόντς. Ε, ξέρω ποια είναι αυτή η δύσκολη μάχη για τον ποιον κατανομάζουμε και ποιον δεν κατανομάζουμε ως ε, οργανισμό και Ινστιτούτο Κατάρτισης. Ε, για το συμβασμό που έχει προταθεί δεν έχω αντίρρηση, αλλά θα το εκτιμούσω ιδιαίτερως αν και άλλα μέρη έχουν τέτοιους ίσους όρους ανταγωνισμού ή ίσο πεδίο, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε τέτοια κατάρτιση. Και εγώ είμαι μέλος ε, της Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά και εκεί πέρα παίζουν και άλλα συμφέροντα. Τώρα, Πρόεδρε, το ζήτημα των ναρκωτικών. Δύο σημεία έχω εδώ να αναφέρω. Είδα ότι και άλλοι συνάδελφοι θέλουν ε, να, να εισαγάγουν τη διαφοροποίηση μεταξύ μαλακών και σκληρών ναρκωτικών. Συμφωνώ εδώ με τον κύριο Κλάς ότι μάλλον αυτό αφορά άλλο πρόγραμμα. Αλλά η διαφοροποίηση, αυτό ο διαχωρισμός ε, μεταξύ μαλακών και σκληρών ναρκωτικών ήδη υφίσταται. Ε, στην Ολλανδία λέμε σχεδόν ότι το χόρτο είναι καλύτερο από την ερωίνη. Επομένω, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ε, μετά, για την υγειονομική περίθαλψη. Ο εκπρόσωπο και το στήμα τη πρόληψη. Ε, ο εκπρόσωπο του Συμβουλίου λέει ότι δεν έχει υπάρξει απόφαση, αλλά εγώ δεν ε, θεωρώ ότι μπορούμε να αποδεχθούμε ε, μια τέτοια κατάσταση και θέλω να μας πούνε ξεκάθαρα ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο αν η πρόληψη και η οικονομική περίθαλψη δεν έχουν θέση σε αυτό το πρόγραμμα τότε πού ακριβώς θα ενταχθούν και πώς μπορούμε ε, να το χειριστούμε από δικαστικής πλευράς. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Συμφωνώ μαζί σας ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσει τα του οίκου του, όμως ε, δεν ε, μπορούμε να αποδεχθούμε και την ε, περιττή γραφειοκρατία. Δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούμε να αποδεχθούμε την προσέγγιση Bellinger και Κλάς σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. We thank you. Ευχαριστούμε για τις δηλώσεις σας, κύριε Βαντεκάμπ και καταγράφουμε φυσικά τη σημασία του θέματος των δημοσιονομικών πόρων που υπογραμμίσατε ιδιαίτερα. Προφανώς το καταγράφω. Η κυρία θα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς εγώ καθυστέρησα να έρθω και δεν μπόρεσα να καταθέσω τροπολογίε σε αυτή την έκθεση που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Αν μπορώ όμω θα ήθελα να σα υποβάλω κάποιε ιδέε που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμε για την Επιτροπή μα και για την μελλοντική συζήτηση για το πρόγραμμα δικαιοσύνη. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι η Επιτροπή μα έχει αντιμετωπίσει το πακέτο δικονομικών εγγυήσεων και στη συνέχεια την έκθεση για τα θύματα που είναι και ένας νέος οδικός χάρτης στην Ευρώπη σε σχέση με την εφαρμογή της δικαιοσύνης. Και όλα αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στο δημοσιονομικό πλαίσιο λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει με τις ε, νέες διαδικασίες δικονομικού χαρακτήρα και την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεύτερον, σε σχέση με τη θέση που μπορεί να έχει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε αυτό το πλαίσιο και εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει εγκάρσιο χαρακτήρα και επηρεάζει πολλά τμήματα του πακέτου, όχι μόνο τις δημόσιες ελευθερίες και όχι μόνο τη δικαιοσύνη, αφορά τα θέματα εσωτερικών, αφορά τα θέματα κοινωνικής αρρωγής και φυσικά επηρεάζει και τα ίδια τα θύματα του εμπορίου ναρκωτικών. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο για την γραμμή κατάρτισης, όπου στη χώρα μου παραδείγματος χάρη υπάρχει μεγάλη έλλειψη για την κατάρτιση εισαγγελέων που να είναι εμπειρογνώμονες στα χρήματα οικονομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσει κανείς να καταδιώξει τα δίκτυα λαθρεμπόρων ναρκωτικού. Και εκεί υπάρχει, όπως σα είπα, ένα πρόβλημα στη χώρα μου για εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν καλά τα χρήματα οικονομικά. Είναι απαραίτητο να διαδραματίσει η δικαιοσύνη σωστά το ρόλο της στην ε, δίωξη του λαθρεμπορίου εγκλήματος. Με την καλύτερη, με την καλύτερη ε, κατάρτιση των δικαστικών, αλλά και μια καλύτερη κατάρτιση διαμεσολαβητών. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στους μικρολαθρεμπόρους ναρκωτικών να αποφύγουν την, ε, τη φυλάκιση εάν ε, δεχθούν να σταματήσουν τις ενεργείες τους. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη βία κατά των ανηλίκων, είναι πολύ πιο δύσκολο να έχει κάνει ένα πρόγραμμα διαμεσολαβητών αλλά τα προγράμματα αυτά μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία και μπορούν να είναι ενδιαφέροντα για όλου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν για τα θέματα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτό το οποίο είναι αρμοδιότητα ε, των ε, δικαστικών αρχών με αυτό που είναι αρμοδιότητα των Υπουργείων Εσωτερικών και αυτό που είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής γιατί η υποστήριξη προς τους τοξικομανείς είναι ένα τέτοιο θέμα Νομίζω ότι η συζήτηση για τα ναρκωτικά και τα εξαρτημένα άτομα δεν έχει καμία σχέση με τον κοινωνικό χώρο και μόνο. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εμπίπτει στον ποινικό κώδικα κάθε χώρας και δεν νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα εδώ. Ο Λουίς Μπέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προσπάθεια των εισηγητών ήταν ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα από τους δύο εισηγητές ενώ. Και στην Επιτροπή Ελευθεριών ε, πράγματι ε, εκτιμούμε το γεγονός ότι μπορούμε να συνεργαζόμαστε σαν δύο επιτροπές, κάτι το οποίο βελτιώνει την νομοθετική μας προσπάθεια, η οποία είναι ιδιαίτερα θετική συμφωνούμε ομόφωνα σε ένα σημείο, ότι θα πρέπει να οικοδομήσουμε το ταχύτερο δυνατόν έναν δικαστικό ευρωπαϊκό χώρο, ένα σύστημα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, το οποίο να είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό. Και τελικά η αρχιτεκτονική της έκθεσης η οποία μας έχει προταθεί και μέσω των τροπολογιών ανταποκρίνεται σε αυτόν τον σφαιρικό στόχο και η πολιτική μου ομάδα είναι υπέρ των τροπολογιών των περισσότερων και ελπίζουμε να καταλήξουμε και στις συμβιβαστικέ. Νομίζω ότι όπως και άλλοι συνάδελφοι θεωρούμε ότι κάτι λιγότερο από 100 τροπολογίες δεν είναι ένδειξη δυναμίας και συνεννόησης, αλλά ε, δείχνει το ενδιαφέρον και τον δυναμισμό των βουλευτών για μια προσπάθεια που αποτελεί θα έλεγα έναν από τους πυλώνες του κοινοτικού δικαίου και της χρήσης του από τους πολίτες. Αυτά είναι σημαντικότατα για τους πολίτες και για αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη από τη δικαιοσύνη και, αυτούς, ε, και για αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται και για αυτούς ε, που βρίσκονται υπό έρευνα. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου και μέσω του αριθμού των τροπολογιών. Μπορείς να μακρηγορήσω, θα ήθελα να επιμείνω σε τρία πιο συγκεκριμένα σημεία πέρα από τα σχόλια, τα οποία ήδη έγιναν, πολύ πλούσια και επικοδομητικά. Το ένα αφορά τα ναρκωτικά και το άλλο κάποιες διακρίσεις, οι οποίες δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξουν στο συγκεκριμένο κείμενο. Χωρίς να επιμείνω λοιπόν, Βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξουν δραστικές δημοσιονομικές περικοπές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να γίνει στη συγκεκριμένο πεδίο και ομόφωνα νομίζω θα δώσουμε τη μάχη για να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική κάλυψη. Τρία επιπλέον συγκεκριμένα σημεία. Επιμένω μέσω των τροπολογιών που κατέθεσε και η ομάδα μου για την βασική εικόνα ορατότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει το πρόγραμμα. Ενθυμίστε ότι στο παρελθόν πολλές δράσεις δεν είχαν προχωρήσει. Με το πρόγραμμα Πανδώρα είχαμε θεωρήσει ότι δεν υπήρχε κατάλληλη υποδομή νομομαθών που να προωθήσουν ακριβώς τα προγράμματα. Δεν είχαν υπάρξει προτάσεις δράσης Πολλές φορές τα κείμενά μας ήταν τόσο δυσνόητα και περίπλοκα που απογοήτευαν όσους θα μπορούσαν να τύχουν τη στήριξή τους. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία το κείμενό μας να είναι εύκολα ορατό, κατανοητό, απλουστευμένο και γι' αυτό ζητάμε να μην αλλάζουν επίσης οι κανόνες από το ένα έτος στο άλλο, να διατηρήσουμε κάτι αναγνώσιμο, προσβάσιμο κάτι το οποίο να εξυπηρετεί πράγματι την υπόθεση την οποία προσπαθεί να προωθήσει η έκθεσή μας. Επίσης και εδώ νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, αν και ίσως να μην ισχύει για όλη την ευρωπαϊκή ζώνη, λέει η ομιλήτρια, όλα τα θέματα της δικαιοσύνης θα πρέπει να είναι στο δίκτυο και διαθέσιμα, προσβάσιμα και κατανοητά. Θα πρέπει δηλαδή εμείς τις γνώσεις των επαγγελματιών να τις προσφέρουμε για χρήση με εύκολο, απλό και σύντομο τρόπο. Λέγεται στο πρόγραμμα της Στοκόλμης κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται εύκολα και πρέπει να το επαναλάβουμε, δεν πρέπει να φοβόμαστε εδώ την επανάληψη, διευκρινίζοντας περί τίνος πρόκειται. Αυτό ήταν το πρώτο συγκεκριμένο σημείο. Το δεύτερο τώρα πάνω στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω. Αφορά μια ευάλωτη κατηγορία, τα παιδιά. Κατέθεσα πολλές τροπολογίες, οι οποίες δεν θέλουν όλες να πούν το ίδιο πράγμα, με πάρα πολύ θετικό τρόπο εγώ Υπογραμμίζω την επιθυμία των δύο συνεισηγητών να προχωρήσουν σε μια συνοπτική, συνθετική και ε, κατανοητή παρουσίαση. μένοντας πάντα στον χώρο του συγκεκριμένου, ιδιαίτερα στην περίπτωση της αντιμετώπισης των προβλημάτων των παιδιών. Νομίζω επίσης ότι η διασύνοριακή συνεργασία θα πρέπει να τύχει πιο ουσιαστικής και συγκεκριμένης στήριξης. Εγώ το ζω αυτό στην περιοχή από την οποία προέρχομαι. Έχουμε πολύ λίγους ε, γείτονες εκεί, τρεις Ευρωπαίους και έναν μη Ευρωπαίο. Τι εννοώ με αυτό, είμαστε θα έλεγα ένα ευρωπαϊκό εργαστήρι και η συνεργασία, τα προγράμματα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και η επιθυμία γενικότερα να υπάρξουν περισσότερες αμοιβαία περισσότερες γνώσεις, κάτι τέτοιο δεν είναι μόνο μέσω οικοδόμησης του δικαστικού χώρου, του χώρου της δικαιοσύνης, του ευρωπαϊκού, αλλά της ίδιας της Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις Πάντως ε, εμείς θα εμείνουμε σε θέματα ουσίας. Σχετικά με τις υπόλοιπες τροπολογίες, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές, οι οποίοι εμένουν σε θέματα όπως η πολυγλωσία. Ε, θα έλεγα θέματα τέτοια τα ξεχνάμε λίγο τον τελευταίο καιρό λέγοντας ότι όλοι θα πρέπει να μιλάμε αγγλικά πλέον αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα ε, είμαι υπέρ αυτού του ευρωπαϊκού χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και η πρόταση που γίνεται. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τους δύο εισήγητες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε και θα το συζητήσουμε και στο επόμενο σημείο της Μεσηδιάδης. Κυρία Αργετίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως ε, δεν θα σας ε, προκαλέσει έκπληξη. Βεβαίως και αναφέρομαι στο θέμα της ε, χρήσης ναρκωτικών, της πρόληψης και καταπολέμησης της. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες για αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά την ε, εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το θέμα, ακριβώς επειδή το θέμα των ναρκωτικών υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα δικαιοσύνης, θα πρέπει να ε, εστιαστεί στην καταπολέμηση της, ε, του εμπορίου ναρκωτικών και άλλων δραστηριοτήτων κατά τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ε, τέτοια προσέγγιση. Οι εγκληματικές δραστηριότητες βεβαίως πρέπει να καταπολεμούνται, αλλά επιστρέφουμε πάντα στη συζήτηση για τα ναρκωτικά. Εάν μπορούμε να τα ε, απαγορεύσουμε ή... Ε, πρέπει κάποια στιγμή να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να μην κάνουν ε, λάθη και αν αυτοί κάνουν λάθη και αποκτήσουν έναν εθισμό πώς θα τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν αυτόν τον εθισμό ή πώς τους βοηθάμε να συνεχίσουν τη ζωή τους αν δεν καταφέρουν να ε, ξεφύγουν από αυτόν τον εθισμό. Τα απαγορεύουμε λοιπόν ή τα ε, διατηρούμε ως ε, συστατικό της κοινωνίας. Αυτό ε, παραμένει ως συζήτηση και βλέπω ότι οι συνάδελφοι ε, έχουν ήδη ε, διαλέξει στρατόπεδο. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει πλειοψηφία για την ε, νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Επομένω, ω συμβασμό, προτείνουμε την διευκόλυνση τη πρόληψη και τον εστιασμό στην διευκόλυνση. Εσείς μιλήσατε για μια διαφοροποίηση μεταξύ μαλακών και σκληρών ναρκωτικών. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Είναι γνωστή η συζήτηση βεβαίως και είναι πράγματι κάποια ναρκωτικά που ε, θεωρούμε μαλακά δεν είναι και τόσο μαλακά τελικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ε, ποινικοποιήσουμε τα πάντα ε, τα οποία προσφέρουν μια ευχαρίστηση στους ανθρώπους. και άλλα είδη ναρκωτικών δεν μπορούμε έτσι απλά να τα ποινικοποιήσουμε. Και δυστυχώς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εάν ε, κάποιοι κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών στον ελεύθερο του χρόνο, αν θέλετε, τότε δεν πρέπει να τους ε, σύρουμε και στα δικαστήρια. Αυτό είναι ο δικός μας φόβος και με αυτό το πνεύμα πρέπει να εξετάσετε τι τροπολογίες Μα Ευχαριστώ. Mrs. now Mr. De Jong, yours is the floor. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις της κυρίας Αργεντίνη. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Ντεκάμπ να πάμε μαζί σινεμά, γιατί ε, ε, θα βγουν δύο ε, καινούργιες ταινίες που δείχνουν πως ε, μία σωστή πολιτική για τα νοκοτικά δεν είναι πάντα κατασταλτική πολιτική. Ε, δεν ε, απαιτείται ποινικοποίηση για όλα τα ναρκωτικά. Θα ήθελα όμως να προειδοποιήσω αυτή την Επιτροπή ε, ότι μπορεί να, μπει σε μια, να πέσει σε μια παγίδα, να κατακαιρματίσουμε όλη αυτή την πολιτική και να ζητήσουμε χρηματοδότηση για όλα αυτά τα σημεία. Εμείς καταφέραμε να, να, προτείνουμε και εξοικονομήσει για κάποια τμήματα αυτής της πολιτικής. Ε, και την εξοικονόμηση λοιπόν θα πρέπει να την έχουμε κατά νου. Για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία βεβαίω πρέπει και να υπάρχει, ε, ιδίως ότι αφορά την ευαισθητοποίηση, το awareness raising, ε, και εκεί τα ίδια κρατημέλη μπορούν να κάνουν πολλά, να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Ε, αυτό ε, είναι κατά το πνεύμα των ε, τροπολογιών μου ότι δηλαδή αυτή η χρήση των ε, δικτών για την μέτρηση των αποτελεσμάτων είναι σημαντικό στοιχείο και θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε και μια παράγραφο στο προήμιο ε, για το γεγονό ότι οι δικαστέ βεβαίω και θα πρέπει να καταρτίζονται, αλλά αυτό δεν χρειάζεται πάντα να γίνεται μέσω εργαστηρίων ή με ανταλλαγέ ε, στι Βρυξέλλε. Αυτό μπορεί να γίνει και σε εθνικό επίπεδο κάλλιστα. Και έτσι θα γίνει η εξοικονόμηση πόρων. Τελευταία παρατήρηση. Διαφωνώ κάθετα με, την, ε, με το να ονομάσουμε εδώ συγκεκριμένε οργανώσεις ή οργανισμού ε, σε ένα κείμενο που είναι πολιτικό, πολιτικό κείμενο αυτού του Κοινοβουλίου, αν εξετάσουμε την ε, ενιαία αγορά και τις αρχές του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Ε, και θα ξεκινήσει μια ολόκληρη διαδικασία αν κατανομάσουμε συγκεκριμένου οργανισμού και όχι άλλου. Γι' αυτό σα καλώ να δούμε μήπω μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ή να, να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα. Ε, και εγώ αναμένω τι συμβαστικέ τροπολογίε ε, και για τα ναρκωτικά και για του δείκτε. Μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, Τσιεύκα για την νομική επιτροπή. Το λέω σωστά. Τσιεύκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι εύκολο συνδυασμό συμφώνων, αλλά εγώ σας θαυμάζω για την προσπάθειά σας. Να επανέλθω σε αυτά που ακούσαμε μόλις. Συζητήσαμε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Διαμακρών θέματα που συνάπτονται με τους στόχους του προγράμματος δικαιοσύνης. Αξίζει να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι. Γιατί η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά μπαίνουμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες και που πρέπει να καλυφθούν από διαφορετικούς κανονισμούς. Ο στόχος του προγράμματος δικαιοσύνης είναι να οικοδομήσουμε ένα κοινό χώρο δικαιοσύνης καλύτερα όπως το είπε ο, ο κ. Μπερλίνγκουερ μια κοινή κουλτούρα μια κοινή δικαστική κουλτούρα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για να φτάσουμε σε εκεί θα πρέπει να προετοιμάσουμε προγράμματα εκπαίδευσης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει αυτό διαφορετικά. Δεν μπορούμε απλώς να διατυπώνουμε και να δημοσιεύουμε έγγραφα στο διαδίκτυο. Θα πρέπει κανείς να μπορεί να τα κατανοήσει, να τα συνδέσει με την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Θέλω να τονίσω λοιπόν το γεγονός ότι τα διαμεθοριακά προγράμματα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την νομ... δικαστική, ενιαία δικαστική κουλτούρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι μετά από την εξέταση των τροπολογιών ότι ξεπενούν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τεγιόγκ. Ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και οργανισμούς οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία για τα θέματα αυτά και να είναι αυτοί οι φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν την κατάρτιση, τα συνέδρια και τις συνδιασκέψεις σε διαμεθοριακό επίπεδο και συγχρόνως θα μας δώσουν μια εγγύηση ότι θα παράσχουν ένα έργο ποιότητος. Και δεν πρέπει εμεί να αυταπατώμεθα χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορεί να καταστεί πραγματικότητα. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα όταν γίνεται κάτι το οποίο είναι θετικό, το οποίο είναι χρήσιμο. Τότε πρέπει να το τονίσουμε και ιδίω πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι ο δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε εάν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε αυτή την ε, δικαστική κουλτούρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μομπάη. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχει σημασία να πούμε ότι όσο τεχνική και αν είναι η προσπάθεια που κάνουμε σε τέτοιους τομείς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ασχολούμεθα με πραγματικούς ανθρώπους με ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές είναι δυστυχείς και υποφέρουν. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι σε μια περίπτωση η οποία έχει σοκάρει την Ουγγαρία και θα ήθελα να συνδέσω τις προτάσεις μου σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται για τον Κίραν Τόιμπιν, έναν Ιρλανδό τραπεζίτη που σκότωσε δύο παιδιά δύο ετών και πέντε ετών σε ένα ατύχημα μια ακραία περίπτωση επικίνδυνης οδήγησης, του ε, επιτράπηκε να επιστρέψει στην Ιρλανδία με αναστολή ουσιαστικά, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση, αλλά δεν έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, ούτε και έχει ε, υπηρετήσει, θα έλεγα, την ποινή του ε, στην Ιρλανδία. Πρέπει να πούμε λοιπόν εδώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα αναλυτών, ερευνητών, οι οποίοι θα ελέγξουν σωστά τις περιπτώσεις ε, δικαστικής συνεργασίας σε τακτική βάση και να καταλήξουν σε συμπεράσματα προτάσεις. Ε, το δεύτερο θέμα είναι η σημασία που έχει η δυνατότητα και η διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων στη δικαιοσύνη. Τμήμα της έλλειψης δικαιοσύνης στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι γονείς των παιδιών αυτών ήθελαν να πάρουν μέρος στις διαδικασίες, στις δικαστικές στην Ιρλανδία, ήθελαν να πάνε στα δικαστήρια, να παρακολουθήσουν τι ακριβώς ε, συμβαίνει εκεί και δεν τους δόθηκε καμία απάντηση στο αίτημά τους, δεν ελήφθη διόλου υπόψη το αίτημά τους. Και ο Ιρλανδός πρέσβης ποτέ δεν απάντησε στις επιστολές που έστειλαν τα δύο αυτά θύματα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πλέον τα συμφέροντα των θυμάτων ή των εκπροσώπων των θυμάτων. Συμπερασματικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να πούμε ότι η πρόσβαση των εκπροσώπων των θυμάτων σε διαμεθοριακό επίπεδο στις διαδικασίες της δικαστικές θα πρέπει να γίνει αντικείμενο εγγύησης και ιδιαίτερα ορισμένες περιπτώσεις αποτυχημένης συνεργασίας δικαστικής, γιατί σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη δεν έφερε εις πέρα στην αποστολή της, δεν τιμωρήθηκε το έγκλημα, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να αναζητηθούν ε, πιο, ε, πιο στεκτικά και θα πρέπει να σας ζητήσω από όλους να βοηθήσετε να υπάρξει δικαιοσύνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επανέρχομαι τώρα στους δύο εισηγητές. Ο κύριος Μπερλίνγκουερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πράγματι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε καταρχάς να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση. Θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση η οποία προηγήθηκε και η οποία έχει ξεκινήσει από την αρχή της διαδικασίας υπογράμμισε την σωστή χρήση του 52 και τη δυνατότητα που δίνουν να συνεργάζονται οι δύο κοινοβουλευτικές ε, επιτροπές. Χαίρομαι εδώ που βλέπω τόσους εραστές της δικαιοσύνης και ε, γενικότερα ε, του δίκαιου στην Ευρώπη γιατί έχουμε την τάση να ασχολούμεθα όλοι με τα οικονομικά κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση αλλά δεν είναι το πάνω η ολοκλήρωση η ευρωπαϊκή περνάει και μέσα από μια κοινή μορφή δικαιοσύνης τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της θα πρέπει να εξυπηρετηθούν και από την δυνατότητα πρόσβαση στη δικαιοσύνη, από την ανταπόκριση της δικαιοσύνης στις προσδοκίες του λαού. Αυτό δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό που ενισχύει την δημοκρατία, αλλά είναι και ένα θα έλεγα χαρακτηριστικό και παράγον της ανάπτυξης. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά στην ανάπτυξη των μορφών συνύπαρξης των Ευρωπαίων. Πολλές από τις τροπολογίες που έχουν ε, παρουσιαστεί και το ενδιαφέρον των συναδέλφων αποδεικνύουν ότι πράγματι εμείς αντιπροσωπεύουμε ένα σημαντικό κομμάτι της Ευρώπης. Να προσθέσω επίσης κάτι άλλο εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπενθύμησε όπως και η σημερινή συζήτηση άλλωστε ότι αν εμείς εμείνουμε σε μια υπερβολική μορφή διακανονιστικής πίεσης τότε φοβάμαι ότι ε, δεν θα έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο απλούστευσης και καλύτερης κατανόησης. Βέβαια δεν πρέπει να είμαστε μόνο πολιτικοί στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και νομομαθείς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς να δεχθούμε τα αιτήματα τα οποία ζητούν μέσω των τροπολογιών στο τελικό κείμενο να υπάρχουν αναφορές σε όλα τα επιπλέον στοιχεία. Παρ' όλα αυτά το τελικό κείμενο θα πρέπει να είναι ένα κείμενο θα έλεγα με σωστή μορφή το οποίο να είναι άμεσα εφαρμόσιμο περιλαμβάνοντας όμως παράλληλα όλα τα επιμέρους μικρότερα στοιχεία όπως έχει ζητηθεί. Γι' αυτό ακριβώς και μέσω της στενής συνεργασίας με τον κύριο Κλάες και με τους Κιώδης θα μπορέσουμε νομίζω εμείς να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα τα οποία ακούστηκαν και τα οποία δεχόμαστε αλλά θα έλεγα χωρίς να μπούμε στη λογική του να πλημμυρίσουμε το κείμενο με λεπτομέρεια. Τώρα κάποια επιπλέον στοιχεία. Πρώτον, το θέμα των θυμάτων. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω, το θέμα αυτό παραμένει στο εσωτερικό του προγράμματος και οφείλεται στο ότι η τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των θυμάτων είναι πλέον μία πραγματικότητα. Στα πλαίσια της δικαστικής παράδοσης τα θύματα δεν ήταν πάντα το βασικό πρόβλημα. Ξέρετε ότι υπάρχουν εγγυήσεις στα πλαίσια των παραδοσιακών μορφών δικαιοσύνης για την υπεράσπιση των ενόχων ή των κατηγορουμένων, αλλά παρόλα αυτά το να μπορέσουμε εμείς να προωθήσουμε κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα και σε διαμεθοριακό επίπεδο, αλλά όχι μόνο για την προστασία των θυμάτων, είναι κάτι το καλό. Ένα άλλο επιμέρους θέμα για το αν θα αναφερθούμε συγκεκριμένα σε αυτούς που μπορεί να, να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό εμείς να προσπαθήσουμε να παράγουμε κανόνες οι οποίοι να μην επικαλύπτονται με προηγούμενες ισχύουσες ρυθμίσεις. Η σχέση λοιπόν ανάμεσα στην αιτιολογική σκέψη και στο επίσημο κείμενο θα πρέπει να είναι μια ε, ισόρροπη σχέση. Εμείς ε, βάλαμε κάποιες αγκυρίσεις σε σχέση με το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα της επαγγελματικής ανάπτυξης αυτών που ασχολούνται με το δίκαιο, με τη δικαιοσύνη, δηλαδή δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι κτλ. Στο πρόγραμμα μας φάνηκε ότι το θέμα αυτό δεν είχε το απαιτούμενο βάρος. Το Κοινοβούλιο τα τελευταία δύο χρόνια πέρασε ορισμένα πολύ σημαντικά ψηφίσματα που προωθούν μία από τις υποθέσεις οι οποίες έχουν γίνει, ότι δεν θα πρέπει να τίνουμε να τα συγκεντρώνουμε όλα, δεν θα πρέπει να τα κάνουμε όλα στις Βρυξέλλες, αλλά και στα κρατημέλη, θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες κατάρτισης, προσπάθειες επιμορφωτικές ε, αυτών που ασχολούνται με την δικαιοσύνη, των επαγγελματιών της δικαιοσύνης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαχυθεί σε όλες τις χώρες μέσω ενός επιτόπου, ενός τοπικού πρωταγωνιστικού ρόλου όλων των εμπλεκομένων την απονομή της δικαιοσύνης και οι οποίοι καλούνται να ανανεώνουν συστηματικά το επαγγελματικό τους νομικό γνωστικό πλωστάσιο. Ευχαριστώ. Κύριε Κλάς για να κλείσει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι βεβαίως και δεν έχω ε, δεν είχα αντίρρηση ούτε έκανα παράπονο για τον αριθμό των τροπολογιών. Απλώς ε, με εξέπληξε ο αριθμό τους. Υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία δεν θα ήθελα να απαντήσω τώρα και με συγχωρείτε γι' αυτό. Σε τρει ε, παρατηρήσει θα περιοριστώ. Πρώτον, για το ύψο του προπολογισμού. Ο κύριος Βαντεκάμπ είπε ότι θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το σημείο. Βεβαίως, παντού αναφερόμαστε στον προπολογισμό Σίγουρα δεν πρέπει να μιλάμε για μειώσει προπολογισμού κτλ. Εδώ μιλάμε για πρόταση. 472 εκατομμύρια ευρώ για την ε, περίοδο 14-20. Εκεί πρέπει να μείνουμε και να μην λέμε τίποτα παραπάνω. Για το level playing field, το ίσο πεδίο ανταγωνισμού, κατά βάση συμφωνώ με αυτή την αρχή. Ο κύριος Δεγιόν ε, έχει εκφράσει ανησυχίες ότι ενδεχομένως και άλλες αρχές ε, θα μπορούσαν να εμπλακούν σε αυτό το θέμα εάν δοθεί εντύπωση ότι κάποιοι οργανισμοί ε, αναφέρονται επί παραδείγματι. Να σας καθησυχάσω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβασμό. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν οπωσδήποτε να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί και κάποιοι όλοι. Ε, εν είδη συμβασμού μπορώ να πω ότι καθαρά ως παραδείγματα να αναφερόμαστε σε τρεις οργανισμούς αλλά ε, στις ε, αιτιολογικές σκέψεις, στο προήμιο και όχι στο διατακτικό. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορώ να ε, διασκεδάσω τις ανησυχίες και των δύο πλευρών. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι στηρίζω ιδιαίτερως ε, τις ε, τροπολογίε όπω κυρία ε, Γκρίσμπερκ για την στήριξη της διαφάνεια και της αναγνωσιμότητας των κειμένων, της προσβασιμότητα των διαδικασιών. Τέτοιες τροπολογίε βεβαίω και τι στηρίζω, όπως και ο συνεισηγητή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλου όλα τα μέλη τα οποία έλαβαν μέρο σε αυτή τη συζήτηση. Κάτι που μα επιτρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη, το σημείο υπαριθμών 5. Προβλέπουμε μισή ώρα για αυτό το σημείο και θα ήθελα να σας παροτρύνω εξ αρχής να το έχετε αυτό υπόψη σας γιατί στις 11 και 10 θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις ε, ψηφοφορίες. Βλέπω όλο και περισσότερα μέλη να προσέρχονται. Σας λέω και πάλι, πρέπει να κλείσουμε σε 30 λεπτά. Να εξετάσουμε λοιπόν τις τροπολογίες στην πρόταση του κανονισμού που θεσπίζει το πρόγραμμα δικαιώματα και ηθαγένεια για το 2014-2020. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κίνγα Γκιόντς και έχει να αντιμετωπίσει 140 τροπολογίες και 45 δικές της. 185 στο σύνολο λοιπόν οι τροπολογίες. Ισχύει και το άρθρο 50 του κανονισμού συνδεόμενες επιτροπές. Επομένως, συμμεριζόμαστε αυτό το φάκελο μαζί με τις επιτροπές ε, γυναικών και απασχόλησης. Αλλά είμαστε η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Θα ακούσουμε και το Συμβούλιο και την Κομισιόν εφόσον θέλουν και εφόσον πρόκειται να το κάνουν εν συντομία και χαιρετίζουμε και τον εισηγητή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τον κύριο Μπόλαντ, ο οποίος είναι παρόν βέβαιος. Καλώς ήλθατε. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια και θα συνεχίσει η συζήτηση. Κύριε σας ευχαριστώ. Είπατε ότι υπήρχαν 140 τροπολογίες που κατατέθηκαν από τα μέλη που καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος και επειδή έχουμε μια κοινή ευθύνη για ορισμένα άρθρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, σειρά τροπολογιών που προήλθαν από την Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών, 51 από την Επιτροπή Απασχόληση και πάνω από 100 από την Επιτροπή Γυναικών. Για το χρονοδιάγραμμα επίσης, <clears throat> η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών θα ψηφίσει σήμερα ή αύριο. Η ΔΕ Επιτροπή ε, Απασχόλησης θα ψηφίσει στις 9 Οκτωβρίου. Επειδή γνωρίζω τις τροπολογίες, νομίζω ότι μπορούμε ήδη να ξεκινήσουμε την επεξεργασία των συμβαστικών λύσεων, γιατί βρισκόμαστε υπό χρόνου όλες οι επιτροπές, μάλλον η δική μας επιτροπή θα πρέπει να έχει τελειώσει τη διαδικασία στις 26 Νοεμβρίου, επομένως πρέπει να προετοιμαστούν οι συμβαστικές προτάσεις και έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές συναντήσεις για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εισηγητών και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις θέσεις των μεν και των δε. Να σας παρουσιάσω λοιπόν μερικά από τα πιο προβληματικά σημεία και τα θέματα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συζητήσεις. Υπήρξαν πολλές τροπολογίες που καλύπτουν τον τομέα της πρόληψης των διακρίσεων, της αντιμετώπισης των διακρίσεων με διαφορετικές διατυπώσεις. Κάποιες χρησιμοποιούν τη διατύπωση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, άλλες χρησιμοποιούν τη διατύπωση της συνθήκης Λισαβόνας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όμως ποια διατύπωση θα προκρίνουμε για να έχουμε μια πιο ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αυτό είναι ένα λοιπόν από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις διαπραγματεύσεις. Ένα περαιτέρω θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι το θέμα των γλωσσών. Είναι από τη μια πλευρά θετικό. Πολλές τροπολογίες τονίζουν ότι οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος, η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να διατυπώνονται σε όλες τις ε, γλώσσες. Βέβαια αυτό τροχοπεδεί και επιβραδύνει τη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τον τρόπο τον πιο αποτελεσματικό για να υπάρχει προσβασιμότητα από τις ΜΚΟ και τους άλλους φορείς που θα είναι τελικοί αποδέκτες αυτών των κονδυλίων, αλλά χωρίς υπερβολική καθυστέρηση. Μια άλλη επίμαχη πλευρά είναι το αν θα είναι εξουσιοδότηση ή εφαρμοστική πράξη που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι ανάλογο με το, τα προβλήματα του προβλήματος του προγράμματος για τη δικαιοσύνη. Τα έχουμε συζητήσει και με τον εισηγητή του προγράμματος δικαιοσύνης. Θέλουμε φυσικά να έχουμε κάποια επιρροή στα ετήσια προγράμματα. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό θα καθυστερήσει η διαδικασία με τον τρόπο αυτό. Είναι όμω απαραίτητο να έχουμε κάποιο έλεγχο για τα θέματα αυτά και νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά επίση. Για το πρόγραμμα δικαιοσύνη αναφέρθηκε ότι υπήρχαν πολλέ τροπολογίε που προτείνουν να υπάρχουν συγκεκριμένοι φορεί οι οποίοι θα είναι οι αποδέκτε των κονδυλίων του προγράμματο και πάλι θα πρέπει να συζητήσουμε αν αυτό είναι ο πιο επωφελή τρόπο για να κινηθούμε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένους φορείς μέσα στην ε, έκθεσή μας. Επίσης να σας αναφέρω ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης εισηγείται είναι η Jean Λάμπερτ, η οποία είναι και μέλος της δικής μας Επιτροπής και μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία μαζί της. Επίσης και με την ε, Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών που είναι η Ρεζίνα μπάστου η συγγήτρια και εκεί μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Αυτά ήθελα να πω και θέλω να ευχαριστήσω όλου αυτού που κατέθεσαν τροπολογίε και του κοιόδη συγγητέ που έχουν εμπλακεί από την αρχή στην επεξεργασία των θεμάτων αυτών και φυσικά και τι ε, οργανώσει τις οργανώσεις των πολιτών με τις οποίες ήρθαμε σε διαβούλευση που ζητήσαν να τροποποιηθεί και ο τίτλος και να συμπεριληφθεί και η έννοια της ισότητας ως σημαντικό στοιχείο αυτού του προγράμματος. Κάτι ακόμα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ηθαγένεια. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, οι αποδέκτες, οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα να μην είναι μονάχα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλοι οι διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο νομίζω ότι θα υπάρξει γενική συνένεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη βοήθειά σας και είμαι σίγουρο ότι θα καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Αγγιόντς. Δύο λεπτά λοιπόν για τους ε, υπόλοιπους ομιλητές, η Κομισιόν και το συμβολικό Κύριε Μισού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εισηγήτρια συνόψε τόσο καλά τις ε, τροπολογίες που έχουμε εξετάσει και τα σημεία που έθιξε είναι ακριβώς τα σημεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού. Ήθελα μόνο να πω ότι η δική μας πρόταση βασίζεται στις συνθήκες. Δεν... Ε, η πρόταση δεν περιορίζεται μόνο στους ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα κοινά και οριζόντια θέματα πρέπει να εξεταστούν σε οριζόντιο επίπεδο. Το μοναδικό πράγμα που κάνει αυτό το πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων ε, των φυσικών προσώπων. Με αυτόν τον γενικό στόχο είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε όλες τις ε, κατάλληλε λύσεις ε, στο τελικό σχέδιο πρόταση. Σας ευχαριστώ, κύριε, κύριε από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά ε, Συμβουλίου και πάλι υπάρχει μια γενική μερική προσέγγιση τη 8η Ιουνίου σε σχέση με την αρχική πρόταση τη Επιτροπή. Η γενική μερική προσέγγιση του Συμβουλίου συμπεριλαμβάνει και τον όρο ισότητα στον τίτλο. Έτσι, δικαιώματα, ισότητα και ηθαγένεια. Ε, προσδιορίζει δραστηριότητες και ενέργειες για την προσταθέμενη αξία την ευρωπαϊκή, διασυνοριακό αντίκτυπο, διασυνορική συνεργασία, διεθνικό αντίκτυπο μάλλον και την ε, ε, διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Στους πιο συγκεκριμένου στόχου, περιλαμβάνει την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των ε, μικρών παιδιών, γυναικών, θυμάτων και ευάλωτων ομάδων ευθυγραμμίζει το πρόγραμμα και, και άλλα προγράμματα υπό το πρόγραμμα καταναλωτών, η ελάχιστη χρηματοδότηση που θα δίδεται μέσω επιχορηγήσεων ε, τίθεται στο 65% τουλάχιστον και στους συγκεκριμένους, τους ειδικούς στόχους προωθούμε την ε, ισότητα μεταξύ άντρων και γυναικών και την ε, θετική αντιμετώπιση των σεξουαλικών προτιμήσεων. θα πρέπει να υπάρχει ε, από κοινού εισαγωγή, ε, συμμετοχή και των ε, μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και το Συμβούλιο έχει θέσει και συγκεκριμένα κριτήρια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος. Η Κυπριακή Προεδρία επιθυμεί να διοργανώσει μια τεχνική συνεδρίαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εναρμονιστούν οι ε, τροπολογίες ε, με την Γενική Μερική Προσέγγιση του Κοινοβουλίου. Κύριε Μπόλαν, εκ μέρου ε, τη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θέλετε να πάρετε το λόγο για δύο λεπτά. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και την δυνατότητα που μου δώσετε να παρακολουθήσω τη συζήτηση και να συμμετάσχω για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα από τη δική μας πλευρά. Εμείς έχουμε βέβαια ανησυχίες ότι η συγχώνευση δύο προγραμμάτων μπορεί να αποδυναμώσει τον αντίκτυπο αυτής της γνωμοδότησης. Παρ' όλα αυτά, από τη δική μας πλευρά, μετά τις συναντήσεις με την Κομισιόν και μετά τις συζητήσεις που έχουν λάβει χώρα μέσα στην ΟΚΕ, Εμείς έχουμε διατυπώσει μια γνωμοδότηση. Αναγνωρίζω την υποστήριξη της εισηγήτριάς σας, την οποία συνάντησα μαζί με άλλους ευρωβουλευτές και όλα αυτά μας επέτρεψαν να καταλήξουμε σε ένα σαφές μήνυμα από την πλευρά της ΟΚΕ. Το μήνυμά μας είναι ότι τα επερχόμενα 7 χρόνια που θα είναι και η διάρκεια του προγράμματος τα δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να παίξουν πρωταρχικό ρόλο σε όλο το έργο και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει ιδιαίτερα να εστιάσουμε στον αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών στις ε, γυναίκες, σε άτομα τα οποία είναι ευάλωτα και το νομοθέτημα το οποίο εξετάζεται σήμερα έχει σαν στόχο να προστατεύσει αυτά τα δικαιώματα και έχει σημαντικό χαρακτήρα το σύνολο των προτάσεων τροποποίησης και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αποδυναμώσουν το αντίκτυπο αυτού του νομοθετήματος για τις γυναίκες και για τις ευάλωτες ομάδες και για όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται υπέρ αυτών των ομάδων του πληθυσμού. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και θέλω να ευχαριστήσω και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας βοήθησαν στη σύνταξη της δικής μας γνωμοδότησης και αν μπορούμε εμείς να σας αρρωγήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο θα το πράξουμε πολύ ευχαριστώ από την πλευρά της ΟΚΕ. Ωραία. Αρχίζει τώρα η συζήτηση. Σας τονίζω και πάλι την ανάγκη να είμαστε σύντομοι και να παραμείνουμε στο χρονικό πλαίσιο. Προτείνω να ακουστούν οι σκιοδησιητές κυρία Αντζελίλη, Βίξτρομ, Λάμπερτ, Ρομέρο Λόπεθ, Αντζελίλη, αν μπορείτε να μιλήσετε μέσα σε δύο λεπτά, γιατί στις 11 πρέπει να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκόντς για την προσπάθεια την οποία έχει κάνει. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες. Υπάρχει όμως μια κοινή γραμμή την οποία συμμεριζόμεθα φυσικά και η οποία έχει σαν στόχο την ενίσχυση των αξιών γύρω από την έννοια της έλλειψης διακρίσεων. Μια έννοια η οποία θα πρέπει να τονιστεί όσο περισσότερο γίνεται στο εσωτερικό αυτού του προγράμματος και υπάρχει και μια συγκεκριμένη αναφορά για τις πλέον ευάλωτες ε, κατηγορίες οι οποίες ε, όπως είναι προφανές έχουν ανάγκη μιας κάποιας ισχυρής προστασίας σε εισαγωγικά. Αναφέρομαι εδώ στις γυναίκες, αναφέρομαι στους ανηλίκους και στις ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο όπως ε, οι ηλικιωμένοι ή και αυτοί που παρουσιάζουν φυσικές αναπηρίες. Συνεπώς λοιπόν εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε και την προοπτική της προστασίας των δύο φύλων, της ισοτιμίας συγγνώμη των δύο φύλων, επί τη βάση της επιτυχούς εμπειρίας του προγράμματος Δάφνη. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόγραμμα αυτό για να προλαβούμε και το πρόβλημα της ε, ε, οικιακής βίας που είναι ένας ξεχωριστός συγκεκριμένος στόχος. Και φυσικά τίθεται εδώ και το θέμα των ανηλίκων, ιδιαίτερα το θέμα της εγκατάλειψης των ανηλίκων, της κακομεταχείρισης των ανηλίκων και όλων των μορφών, εν πάση περιπτώσει, παράνομης εκμετάλλευσης και κατάχρηστικής συμπεριφοράς. Έχει σημασία να συμπεριλάβουμε στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλες τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Ευχαριστώ, κυρία Βίξτρομ. Σεσίλια. Time to use the floor. I am so... Χίλια, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Είχαμε μια πολύ ε, ενδιαφέρουσα διμερή συζήτηση με τον συνάδελφο. Καλό θα ήταν και άλλοι συνάδελφοι να το δοκιμάσουμε βεβαίω. Κάποιε φορέ έχει καλά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, ήμουν σκιώδη συγγήτρια από την ομάδα Άλντε και θέλω να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο και ιδιαίτερο στην ευαισθησία και γενεοδορία που έδειξε απέναντι στους συναδέλφους ε, από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, γιατί αυτό καθιστά το έργο πολύ πιο ενδιαφέρον. Η πρόταση της ε, Επιτροπής ε, ε, είναι μια ανάμειξη των διαφόρων ε, προγραμμάτων, αλλά βεβαίως μπορούν να υπάρξουν ε, πολλές βελτιώσεις. Είναι σημαντικό όλα τα μέρη να λάβουν την προσοχή που τους αξίζει. Γι' αυτό και έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Εγώ ανησυχώ ότι, το... ότι δεν θα εστιαστούμε αρκετά στην ισότητα χαιρετήσω τι τροπολογίε ε, για την ε, μεταβολή του άρθρου 4 για του ειδικού ε, στόχους. Είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός των στόχων και υπάρχει ο κίνδυνος ε, αλληλεπικάλυψης και γι' αυτό θα πρέπει να, να χειριστούμε ξεχωριστά τον κάθε στόχο για να ελάβει ο κάθε στόχος την προσοχή που του αξίζει. Θέλω να προσθεθεί και η ξενοφοβία στους στόχους. Εφόσον η ξενοφοβία είναι κάτι που αποτελεί μεγάλο πρόβλημα σε αρκετά κράτη-μέλη και έχουμε δει τρομερά παραδείγματα για τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει και αποτελεί και απειλή για τις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονίσουμε και την ξενοφοβία. Κάτι άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω θα ήταν η σημασία της προώθησης, προστασίας και παρακολούθησης των δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να ε, γινόταν ανέκαθεν, αλλά δεν είναι ποτέ αργά. Επιπλέον, ε, θέλω να εστιαστώ και στην καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ των φίλων, βάση φύλου, αλλά και διακρίσεις που προκύπτουν από, ε, από το φίλο ενός προσώπου. πρέπει πάντα να προωθούμε και να στηρίζουμε το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ε, ε, ασχολούνται σε αυτόν, με αυτόν τον τομέα, γιατί δεν είναι εύκολο για πολλούς, πολλές αυτές τις οργανώσεις. Τέλος, ό,τι και να κάνουμε σε αυτή την έκθεση δεν θα έχει σημασία, εκτός και αν υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση για την κάλυψη των ε, έργων αυτού του προγράμματος. Πρέπει λοιπόν να μερευνήσουμε τόσο ώστε να υπάρχουν επαρκή επίπεδα προπολογισμού για το πρόγραμμα. Η προσέγγιση της συγγήτριας είναι πολύ καλή. Μπορούμε να τη στηρίξουμε εκ μέρους της ε, ομάδας μου και υπάρχουν και προσθήκες από προτείνονται στις τροπολογίες που θα μπορέσουμε να τις συζητήσουμε με τους ε, σκιώδεις. Και ο γενικός ε, στόχος είναι η διασφάλιση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ, κυρία Λάμπερτ. Δύο λεπτά αν μπορείτε. Σα ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κίνγκα Γκένς για την πολύ καλή συνεργασία που επέδειξε με όλους τους σκιοδησιητές. Το θέμα αυτό το επεξεργαζόμαστε και στην Επιτροπή Απασχόληση και προσπαθούμε να βρούμε κάποια συνέργεια μεταξύ των δύο επιτρόπων με στόχο να κατευθυνόμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Να η σημασία της αλλαγής του τίτλου είναι κάτι το οποίο όλοι το χαιρετίζουμε. Νομίζω ότι αντανακλάμε τον τρόπο αυτό καλύτερα το περιεχόμενο του προγράμματος και είμαι σίγουρη ότι για τα θέματα προστασία προσωπικών δεδομένων που είναι ένα από τα θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πρόγραμμα αυτό θα μπορέσουμε επίσης να βρούμε ικανοποιητικές συμβιβαστικέ λύσεις μεταξύ μας. Θέλω να επικροτήσω αυτά τα οποία έχουν λεχθεί και από τους άλλους σχεδόντες εισηγητές, αλλά έχω ένα ερώτημα για το θέμα των δικαιωμάτων των καταναλωτών και του πώς θα συναρμοστεί αυτό με το συνολικό πακέτο. Γιατί πιστεύω ότι για πολλούς από εμά δεν είναι ακριβώς η ίδια κατεύθυνση που ακολουθεί αυτό το θέμα όπως για άλλα ζητήματα που μας απασχολούν που συμπεριλαμβάνει παραδείγματο χάρη στοιχεία του προγράμματο Δάφνη. Είναι λοιπόν αυτό ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα να έχω περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση του. Δύο λεπτά για την κυρία Ρομέρο. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στη φιλοσοφία που διατρέχει το πρόγραμμα αυτό για τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πολλές φορές με το πρόσχημα της απλοποίησης μερικές φορές αφήνουμε κατά μέρος τις προτεραιότητες. Η επικεφαλίδα αυτή που αφορά το, το πρόγραμμα αυτό για το, στο πρόγραμμα αυτό σε σχέση με την πρόληψη της τοξικομανίας νομίζω ότι αφαιρεί και ένα τμήμα των κονδυλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα κατά της βίας. Το πρόγραμμα Δάφνη δεν έχει καμία αύξηση κονδυλίων από το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο σε αυτό το πλαίσιο, όταν έχουμε τονίσει ιδιαίτερα πόσο σημαντική είναι η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Γιατί είναι ένα αδίκημα, θεωρείται αδίκημα σε όλου του ποινικού κώδικε. Αλλά η πρόληψη τη τοξικομανίας είναι ένα θέμα που είναι σε συζήτηση τα ελαφρά ναρκωτικά και τα βαριά ναρκωτικά, αν πρέπει τα πρώτα να αποποινικοποιηθούν κτλ. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στο τωρινό πρόγραμμα. Θα ήταν πολύ πιο λογικό να το αντιμετωπίσουμε σε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία και τι τις κοινωνικές Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν, αν συγκρίνουμε το πόσα πολλά χρήματα δίνονται για την για κατασταλτικές ενέργειες είναι τεράστια τα κονδύλια αυτά σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών που είναι ένα πολύ μικρό ποσό σε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι αλλάζουμε τις ισορροπίες. Το πρόγραμμα για τα εσωτερικά θέματα αντιμετωπίζει περίπου παίρνει ουσιαστικά το σύνολο των κονδυλίων και το πρόγραμμα Δάφνη μένει μονάχα με ένα τα 100 του συνολικού χρηματοδοτικού ε, πλαισίου που έχουμε. Τα υπόλοιπα τα παίρνει το τα παίρνουν τα εσωτερικά θέματα. Λοιπόν, επανέρχομαι στην συγγήτρια μας την κυρία Γκάλ. <clears throat> κυρία Γκρέντς, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι έχετε εκφράσει τις κύριες ανησυχίες που συνάπτονται με αυτό το πρόγραμμα. Από τη μία πλευρά δεχόμαστε την ιδέα ότι διαδέχεται το προηγούμενο πρόγραμμα ή τα προηγούμενα προγράμματα. Αυτό είναι θετικό αλλά οδηγεί και σε κάποιες δυσκολίες. Το θέμα είναι οι στόχοι των προγραμμάτων προ... προηγουμένων προγραμμάτων μπορούν να καλυφθούν με τους διαθέσιμους στόχους. Δεν μιλάω για την Ευρώπη των πολιτών, μιλάω για τους πόρους σε δημοσιονομικό επίπεδο που δεν είναι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ορατή. Αν συγκρίνουμε τους προηγούμενους προπολογισμού για τα τρία προηγούμενα προγράμματα και τον τωρινό προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση χρηματοδοτικών πόρων. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να προκύψει μια πραγματική συζήτηση μεταξύ μας για τον τρόπο με τον οποίο θα καταλήξουμε στις βέλτιστες συμβαστικές λύσεις ώστε να εξυπηρετήσουμε τους στόχους που θέλουμε, όχι να έχουμε υπερβολικό αριθμό στόχων χωρίς επαρκείς πόρους, αλλά συγχρόνως να μην παραλείψουμε τίποτα από αυτά που είναι σημαντικά, όπως παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα Δάφνη, ή όλους τους στόχους, τους νέους στόχους οι οποίοι έλκονται από τις νέες πολιτικές που έχουν διατυπωθεί από την Επιτροπή μας. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε μια συμφωνία πριν περατώσουμε τις διαπραγματεύσεις μας και με το Συμβούλιο. Κατά τα άλλα μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει κάτι ακόμα που ανέφερε η Jean Lambert, το θέμα των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η προστασία των καταναλωτών σε αυτά υπάρχει ένα άλλο ταμείο που καλύπτει άλλες πλευρές της προστασίας των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν και εκεί να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο είναι αποδεκτό και το οποίο συμβάλλει στο πρόγραμμά μας και όχι να υπάρξει σύγχυση μεταξύ των δύο διαφορετικών προγραμμάτων. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν και σας ευχαριστώ και πάλι για τη βοήθειά σας και την ε, υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκόγκ. Τώρα θα θέσουμε την ημερομηνία για την ψηφοφορία προσανατολισμού. Θα λάβει η χώρα στι 26 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Επομένω, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη μέση διάταξη για το επόμενο μισάωρο. Σα υπενθυμίζω ότι έχουμε ε, ψηφοφορία στι 11 και 10. Έχουμε λοιπόν μισή ώρα για το σημείο 6 για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες για την περίοδο 2014-2020. Συνάδελφος ε, Σάμπα Σόγκορ είναι ο εισηγητής. Θα εξετάσουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησής του και μετά για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών. Αυτό θα γίνει στη συνέχεια όμω. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σόγκορ και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη. Να σας υπενθυμίσω ότι ε, για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής ε, Πολιτισμού εδώ μοιραζόμαστε την αρμοδιότητα ε, με αυτή την Επιτροπή. Η καταληκτική προθεσμία είναι πιο σύντομη από αυτό που προβλεπόταν αρχικά. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον εισηγητή και μετά στους υπόλοιπους. Κύριε Σόγκορ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ στενό το χρονοδιάγραμμα πράγματι αυτή η γνωμοδότηση και γιατί η Επιτροπή Πολιτισμού δεν μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία με το Συμβούλιο για τη νομική βάση. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου κατόπιν αιτήματο τη Επιτροπή Πολιτισμού ε, στην γνωμοδότησή της ανέφερε ότι το πρόγραμμα ακολουθεί με έναν διτό στόχο ε, ε, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ιστορία αλλά και την συμμετοχή των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κανένας από τους δύο αυτούς στόχους δεν ε, είναι υποδέστερο του άλλου. Η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διπλή νομική βάση για την υιοθέτηση της πρότασης είναι απαραίτητη. Ε, η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου διαφέρει από αυτή της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου σε δύο σημεία. Πρώτον, ε, αφήνει στον νομοθέτη να αποφασίσει αν οι δύο στόχοι που οι δύο παραπάνω στόχοι πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμοι και ισάξιοι... ή αν ε, ο πρώτος στόχος ε, αφορά την συμμετοχή των πολιτών. Δεύτερον, ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή θεωρούν ότι ο συνδυασμός των άρθρων 3, το 352 και 167 είναι δυνατή. Βεβαίω, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο αυτέ οι δύο διαδικασίε είναι συμβατέ. Μάλιστα, αυτή η γνωμοδότηση, εισάγοντα τον όρο spirit, πνεύμα, γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν. Ε, το remembrance, αυτή η ανάμνηση, το, Νημονικό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής Ταυτότητα, γι' αυτό και ε, με την ε, εισαγωγή αυτή της διάσταση του πνεύματος ε, σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή. Η εισαγωγή της έκφρασης του ευρωπαϊκού πνεύματος σε αυτό το πρόγραμμα για τους Ευρωπαίους πολίτες θα ενισχύσει την προγραμματισμό και υλοποίηση των προϋπολογισμών Ε, και θα προωθήσει τα διεθνή προγράμματα εταιρική σχέση. Αν δεν υπάρχουν φυσικά σύνορα και μοιραζόμαστε τον ευρωπαϊκό χώρο με ε, με τις που παρουσιάζει το ευρωπαϊκό πεδίο θα ε, συνεχίσουμε στον καλό δρόμο που έχουμε χαράξει τα τελευταία 50 χρόνια. Και έχουμε 229 εκατομμύρια στη διευθυνσία μας για αυτό το πρόγραμμα. Και βεβαίως, όπως αναφέρατε, η προθεσμία είναι 26 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Θα, θα δώσουμε τώρα το λόγο ε, στους συναδέλφους. Κυρία Γερόκα, έχετε το λόγο. Ε, what... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω στο σημείο αυτό έσβησε. Η πρόταση της Κομισιόν να θέσει τους Ρωμά στο προσκήνιο των ομάδων εστίασης για το θέμα της ε, υπηκότητας και των στόχων της υπηκότητας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι η Επιτροπή μας αγωνίστηκε υπέρ αυτής της στρατηγικής για τους Ρωμά. Οι πολίτες αυτοί οι οποίοι παραμένουν στο περιθώριο οικονομικά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες να μπορέσουν να ασκήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εγώ θα ήθελα να συμβάλλω στο κείμενο να τονίσω την απαραίτητο να διατηρήσουμε την σημασία της παρέμβασης για αυτές τις ομάδες εστίασης όπως είναι η Ρωμά στις τοπικές κοινωνίες και να τονίσουμε τη σημασία του πνεύματος της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας <clears throat> που προς το παρόν είναι απλώς ένα σχέδιο για το μέλλον. Για μένα σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να υπάρξει η μεγαλύτερη παρέμβαση. Καταρχήν ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγέλς, ως και οδησίητε σας ευχαριστώ και εγώ για το σχόλιο σε σχέση με την νομική βάση. Ελπίζω ότι αυτή η διπλή νομική βάση θα γίνει δεκτή, γιατί αυτό είναι ένα από τα κέρια θέματα. Εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω, γιατί μιλάμε για μια Ευρώπη πολιτών, και όταν μιλάμε για προγράμματα χρηματοδότησης για τους ε, πολίτες και την ηθαγένεια και την βελτίωση της συνειδητοποίησης για την ευρωπαϊκή ταυτότητά μας. Πιστεύω ότι όλα υποστηρίχτούν και σίγουρα αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Εμείς έχουμε εκφράσει τις διαμαρτυρίες μας για τον ευρωσκεπτικισμό, για την χαμηλή προσέλευση των ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές, την ε, το χαμηλό επίπεδο υποστήριξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά θέματα. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε ένα ισχυρό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει σώμα, Ρώμα, περιλαμβάνει τα άτομα τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, την άσκηση των δικαιωμάτων του. και επομένω να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να καταδείξουμε τη σημασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε καθημερινό επίπεδο, πώ μπορούμε να έχουμε ένα αντίκτυπο στου πολίτε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ελπίδα μου λοιπόν ότι μπορούμε από κοινού να αποδειχθούμε αρκετά ικανοί στον αγώνα μας για το πρόγραμμα αυτό και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστούμε, Η κυρία Ρομέρο, Λόπες Ρομέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι σημαντικό αυτό το πρόγραμμα παρά το γεγονό ότι δυστυχώ η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη, όπω είπε και η κυρία Γκιόντ, είναι ανησυχητική. Και δεν ξέρουμε επομένω αν αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσει πράγματι να επιτύχει τους στόχους του. Εγώ πάντως θέλω να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου γιατί πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό έχει μια αποτελεσματικότητα παρά το γεγονός ότι δεν επαρκείς η χρηματοδότησή του. Όπως είπε ο εισηγητής, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το τι σημαίνει η ιστορική μνήμη της συμμετοχής. Πρέπει λοιπόν η συμμετοχή των πολιτών να βασίζεται στις ιστορικές μας μνήμες. Επομένως θα πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο αυτά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η άποψη του εισηγητή. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό να σκεφτούμε τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο τη μειονότητα των Ρωμά που είναι πολύ σημαντική, αλλά και τους μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς που έρχονται στην Ευρωπαϊκή, αποκτούν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, είναι πολύ σημαντικό για όλους αυτούς να κατανοήσουν τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε ιδιαίτερα στα θέματα των μειονοτήτων και να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση και επίγνωση της σημασίας της ε, παρουσίας τους. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση γιατί αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση δεδομένη τη ε, σημασία του. Σα ευχαριστώ κύριε Μάκιντάερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμένα με προβληματίζει πολύ ε, το όλο σκεπτικό του προγράμματος. Ε, πρώτα απ' όλα ανησυχώ για το γεγονός ότι προτείνουμε να, να ξοδέψουμε 229 εκατομμύρια ευρώ ε, στην ε, πρότασή μας για την αύξηση της ολοκλήρωσης, της ενσωμάτωσης. Ε, δεν με χαροποιεί το γεγονός ότι προωθούμε την ε, μεγαλύτερη συνεργασία και στενότερη συνεργασία. Βλέπω και εκτιμώ το γεγονό ότι ο, ο Μπαρόσο μα λέει ότι θέλουμε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Εγώ βεβαίω δεν θέλω ομοσπονδιακή Ευρώπη. Μάλλον πρόκειται εδώ για προπαγάνδα παρά για ε, παροχή πληροφοριών. Δεν θέλουμε να πείσουμε με του πολίτε να ψηφίσουν, που είναι σημαντικό για όλε τι εκλογέ. Πάμε πολύ παραπέρα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει έτσι να ξοδεύουμε τα χρήματα φορολογουμένων. Okay, Ευχαριστούμε κύριε Μακεντάιρ. Κύριε Σόγκορ, κάποιες ε, καταληκτικές παρατηρήσεις. Και να μας πείτε και τι συμβαίνει με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στην κυρία Μακεντάιρ. Αν εξετάσετε το άρθρο για την δομή του προγράμματος και τις υποστηρικτικές ε, ε, ενέργειες. Ε, δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα για την ομοσπονδιοποίηση, που ανέφερε ο κύριος Μπαρόσο. Ουσιαστικά μιλάμε για το για το ευρωπαϊκό πνεύμα και για το πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συναντηθούν, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν τις πολιτιστικές τους αξίες. Δεν νομίζω ότι αυτά τα χρήματα ε, θα σπαταληθούν για την διαμόρφωση ενός ομοσπονδιακού κράτους. Και βεβαίως ελπίζουμε η Επιτροπή Πολιτισμού να καταλήξει σε μια συμφωνία ε, με το Συμβούλιο για το θέμα της νομικής βάσης σε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα και πάλι. Ευχαριστώ. Then, as... Όπως είπαμε εξ αρχής, Υπάρχει προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 26 Σεπτεμβρίου. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε τέσσερα θέματα από τις 11 και 10 και μετά. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Προτείνω να κάνουμε διάλειμμα εφόσον τα καταφέραμε. και για να περιμένουμε κατά μέλη που έχουν προγραμματίσει να βρίσκονται εδώ στις 11 και 10. Γιατί μπορεί να έρθουν λίγο αργότερα. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα 20 λεπτών και επαναρχόμαστε στις 11 και 10.